Eh, eh, Καλημέρα συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Eh, Δεν είναι πολλοί παρόντες. Αυτό διότι υπάρχει ταυτόχρονα μια αντιπροσωπεία εις Λιθουανίαν που θα επισκεφθεί το πυρηνικό, πυρηνικό αντιδραστήρα εκεί. Η κυρία Γιάλα Σέντερ δεν είναι ακόμα εδώ, αλλά θα καταφτάσει όπου να είναι. Οπότε, ε, το σημείο της είναι το σημείο 7, απαλλαγή του Συμβουλίου. Και μετά, το σημείο 12 της κυρίας Ολμάιερ, άμεσες πληρωμές. Κυρία Ολμάιερ, είσαστε εισηγήτρια και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη και συνοπτική. Είναι η γνωμοδότηση για τις άμεσες πληρωμές και παρουσίαση του θέματο στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Και από του στόχου σημαντικότερου τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού πάντα ήταν ο εξή. Από την μία πλευρά θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια και τη σαφήνεια και ταυτόχρονα σε σχέση με το θέμα θέλουμε να μειώσουμε το διοικητικό άχθο για του δικαιούχου και για τα κράτη-μέλη. Ένα λοιπόν από τα σημαντικότερα καθήκοντα και στόχο τη κοινή αγροτική πολιτική μεταρρύθμιση αυτή είναι η μείωση του διοικητικού άχθους για τους δικαιούχους και τα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε το ότι έχουμε σαφή κριτήρια όσον αφορά τη διαφάνεια. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, σε σχέση με αυτό, όσον αφορά τους δραστήριους, ε, τους ενεργούς γεωργούς, το πρασίνισμα της ΚΑΠ, τους μικρούς γεωργούς, ε, και κατεξισοδότηση πράξη που προβλέπονται για όλα αυτά τα θέματα, έχω προτείνει σχετικέ τροπολογίε Και όσον αφορά τι κατεξισοδότηση πράξη για να εξασφαλίσουμε ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είπα ότι δεν θα έπρεπε εμεί εδώ να δώσουμε πολλέ τροπολογίε, όμω έχει προβλέψει πολλέ κατεξοδότητε συμπράξει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το θέμα αυτό των κατεξοδότητων συμπράξεων δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να αφορά, να αφορά την πολιτική ουσία κανονικά αφορά την εφαρμογή ε, ενό θέματο που είναι συμπεφωνημένο σε πολιτικό επίπεδο. Προτείνω λοιπόν διαγραφή κάποιων κατεξουσιοδότησης πράξεων και στις εξηγήσει μου κατέστα σαφέ ότι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή πραγματικά θα έπρεπε να εξασφαλίσει το ότι όλη η πολιτική ουσία βρίσκεται στην βασική πράξη, στο βασικό κείμενο. Ε, σε σχέση με αυτό, όσον αφορά τη διαφάνεια, την απλούστευση και τη μείωση της γραφειοκρατίας, πρότεινα μεταξύ άλλων ότι οι ενεργοί γεωργοί θα πρέπει να καθορίζονται μέσω ενός αρνητικού ε, καταλόγου, να δουν ποιος δεν είναι γεωργός. Να σταματήσει δηλαδή ε, το ανώτατο κατόφλι γιατί αυτό είναι υπερβολική, υπερβολικός διοικητικός ε, φόρτος. Υπάρχουν κάποιες ειδικές διατάξεις σχετικά με την οικολογική διάσταξη, διάσταση και με τις κυρώσεις. Έχει να κάνει με, τις, την πολιτική διάσταση γιατί γνωρίζουμε ότι εντός της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και αυτό ε, είναι ε, σε δημοκρατικό επίπεδο πολύ ε, πολύπλοκο. Ε, επίσης, ε, οι νέοι ε, γεωργοί, θελοντική ρύθμιση, ανάλογα με την ανάγκη των κρατών, θα δούμε πώς θα δημιουργηθεί αυτό το εθελούσιο καθεστώς και όταν κάποιος κάνει ένα αίτημα, θα πρέπει το ίδιο αίτημα να, ε, μην χρειάζεται να ξαναγίνει το επόμενο έτος όταν είναι ίδιο για να μειωθεί έτσι το κόστος. Αυτά γενικά. Ε, χαίρομαι που θα γίνει κάποια συζήτηση και να πω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 12 ε, Ιουλίου στις 12 και γι' αυτό ε, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε με τους συναδέλφους ε, και να πω ότι τώρα είμαι έτοιμη να δώσω το λόγο στο Πρόεδρο. Ehm, Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είδα ότι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα αυτό δεν είχαν έρθει ακόμα. Συγγνώμη γι' αυτό. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα πάρουν το λόγο σχετικά με αυτά που ακούστηκαν από την εισηγήτρια. Υπάρχουν τυχόν σχόλια. Κανένα σχόλιο. Καλώς θα ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο. Όταν οι συνάδελφοι όμως της Επιτροπής, οι ειδικοί συνάδελφοι καταφτάσουν, θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουν αυτά που είπε η κυρία Βολμάιερ. Ζητώ συγγνώμη για μια ακόμη φορά. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο για την ώρα. Περιμένουμε κάποια σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αργότερα. Πάμε στο θέμα που δεν ασχοληθήκαμε χθε. το σημείο 7. Απαλλαγή για το Συμβούλιο. Είναι μακριά ιστορία αυτή, παλιά ιστορία, το θέμα αυτό της απαλλαγής. Νομίζω λοιπόν, κυρία Γιάλα Σέντερ, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι όλη κατάσταση και τι μπορούμε να περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπήρχε κίνηση, συγγνώμη και άργησα να φτάσω. Τέλο πάντων, υπήρχε ένα χάο κυκλοφοριακό. Όπω πολύ σωστά είπατε και εσεί, Πρόεδρε, πρόκειται για μακριά ιστορία. Στο Κοινοβούλιο όμως, όπως και να έχει, συνεχίσουμε να εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον μας, γιατί θέλουμε να εξομαλυνθεί η κατάσταση γιατί φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι τώρα, κατά το παρελθόν, ήταν τα πράγματα ομαλοποιημένα. Σε σχέση λοιπόν με τη χωρίση τη απαλλαγή, θέλουμε το Κοινοβούλιο να είναι πλήρω αναγνωρισμένο και όλα τα θεσμικά όργανα που μέχρι τώρα δέχτηκαν να υποβληθούν στο δημοκρατικό έλεγχο, το έχουν κάνει με εξαίρεση το Συμβούλιο που παρότι διαστόματος πολλών προεδριών έχει πει ότι Βούλετε να ρυθμίσει την όλη κατάσταση, μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει αποκρισταλωθεί. Με ποιο τρόπο δηλαδή θα γίνει. Όχι απλά ο διάλογος, αλλά θα αναγνωριστεί και το δικαίωμα του Κοινοβουλίου. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε επιτύχει. Η νέα πρόταση, επειδή αυτό που κάναμε το Μάιο τελικά ήταν ακριβώς να αναβάλουμε, περιμένοντας ότι η Δανική Προεδρία που είχε δείξει πολύ θετική στάση και πολύ καλές προθέσεις ε, και διάθεση να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια βελτίωση, δηλαδή η Ιδανική Προεδρία να ανταποκριθεί στα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, τώρα έχουμε μια νέα Προεδρία. Έχουμε λοιπόν και μια νέα πρόταση. σε αυτή τη δεύτερη φάση απαλλαγής των ε, θεσμικών οργάνων. Στόχος μας είναι να δούμε τι νέο έχει προκύψει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου δηλαδή και στο πρώτο και στο τρίτο τμήμα. Δικαίωμα του Κοινοβουλίου δηλαδή να δίνει έγκριση και μετά εντοπίζουμε διάφορα σημεία και εμβαθύνουμε σε κάποια από αυτά. Επίσης έχουμε και την αγνομοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου σε σχέση με τα κτίρια υπήρχαν κάποια ανησυχητικά στοιχεία και το Συμβούλιο πολλές φορές έχει πει ότι λαμβάνει υπόψη του τι ε, απόψει του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχουμε λοιπόν στην δική μας πρόταση συμπεριλάβει, συμπεριλάβει κάποια στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι δεν έχει λάβει ακόμη υπαρκώς υπόψη του το Συμβούλιο και αναφέρουμε κάποιες πτυχές που θα πρέπει να βελτιωθούν. Κάποιες από αυτές τις δέχεται το Συμβούλιο, κάποιες άλλες όχι. Αναφέρουμε επίσης και μια σειρά εκκρεμών ε, ζητημάτων. 26 ερωτήσεις είχαν τεθεί στο Συμβούλιο το Μάιο, δεν έχει απαντήσει. Υπάρχει μία μικρή χειρονομία, έστειλαν κάποια κείμενα, τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν απάντηση στα ερωτήματα του Κοινοβουλίου, ούτε καν πρόκειται για τα έγγραφα τα οποία είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά από διαβούλευση και με τους συναδέλφους αποφάσισα να επαναλάβω και κάποιους όρους ε, που είχαμε συμπεριλάβει για να βρούμε μια συμφωνία, μια συνεννόηση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και είναι κάποια θέματα που θα δούμε και στο πλαίσιο του σεμιναρίου για τις διάφορες αρμοδιότητες Συμβουλίου Κοινοβουλίου στον τομέα της απαλλαγής. Είναι κάτι που έχει προτείνει η δική μας Επιτροπή και νομίζω ότι μπορεί να είναι και μια ευκαιρία και να ενημερωθεί η νέα Προεδρία, η Κυπριακή Προεδρία, που μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κάποια αρχικά δείγματα ότι ενδιαφέρεται για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Με τον κύριο Τόιρερ όμω ε, θα προσπαθήσουμε εκ νέου να έλθουμε σε επαφή με τους Κυπρίους για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και φυσικά και θα ακούσουμε τις προτάσεις τροπολογίας και όλες τους, τις άλλες προτάσεις. Θέλω να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως ε, την ε, γραμματεία γιατί χωρίς την πολύτιμη βοήθειά της δεν θα είχε γίνει τίποτε από όλα αυτά και ιδίω για τη μεγάλη υπομονή που έχει επιδείξει η γραμματεία. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο πάνω σε αυτό το θέμα. Σέντεργαρντ, άλλος. Κελακάκης. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας για την καλή δουλειά που έκανε πάνω σε αυτό το θέμα. Ακαθόδες ζήτημα και νομίζω ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η θέση του Κοινοβουλίου μέχρι ότου να υπάρξει σημαντική κίνηση από πλευρά Συμβουλίου. Η ακρόαση είναι μια καλή ιδέα. Μπορούμε να κινητοποιήσουμε και την Κυπριακή Προεδρία, η οποία ενδεχομένως μπορεί να είναι πιο ευέλικτη από ότι πρώτερες προεδρίες και θέλει να πετύχει πράγματα και συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε διαφανείς όσον αφορά τα δικά μας θέματα, τα δικά μας ζητήματα, ανεξάρτητα από αυτά που θέλει ή δεν θέλει το Συμβούλιο. Όπως το λέμε στην έκθεση, εγώ θα ήθελα να δείχνουμε ότι εμείς είμαστε διαφανείς όσον αφορά τα λογιστικά μας, όπως κάθε θεσμικό όργανο θα έπρεπε να είναι. Κάθε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Και βέβαια θα πρέπει να αναβάλουμε τη χορήγηση της απαλλαγής σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την πρότασή της. Έχω τρία θέματα που θέλω να θίξω. Πρώτα απ' όλα, τι μπορούμε να αναμένουμε από την Κυπριακή Προεδρία. Νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να δημιουργηθεί μια κατάσταση κατά την οποία η Κυπριακή Προεδρία με το λίγο χρόνο που απομένει να αλλάξει τη γνώμη του Συμβουλίου. Ας μην τρέφουμε αυτά πάτες. Θα πρέπει να το δούμε σαν μια μάχη μακράς διαρκείας, μακρά διαδικασία. Είναι καλό το να διεξαχθεί μια ακρόαση με τη συμμετοχή της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά ας μην έχουμε αυταπάτες. Η Κυπριακή Προεδρία έχει πολλά άλλα προβλήματα και δεν πρόκειται ξαφνικά ε, να λύσει αυτό το πρόβλημα ε, και να αλλάξει την άποψη της πλειοψηφίας του Συμβουλίου. Αυτό που νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι να ε, την υποστηρίξουμε την Προεδρία, να στείλουμε μια πρόσκληση προς την Κυπριακή Προεδρία όταν θα ασχοληθούμε και θα συζητήσουμε την έκθεση εδώ στην Επιτροπή μας, ούτω ώστε η Προεδρία να μπορεί να συμμετάσχει στη συζήτηση και προφανώς η Προεδρία θα πρέπει να έχει άλλη μια πρόσκληση όταν θα κινηθεί το θέμα στο Κοινοβούλιο. Να είναι σαφές ότι τους προσκαλούμε, γιατί υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες στο Συμβούλιο. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν κάποια μεταφραστικά σφάλματα στο δανεικό κείμενο. Παρακαλώ ας ελέγξουμε λοιπόν τα διάφορα κείμενα, τις διάφορες μεταφράσεις και να εξαφανιστούν τα μεταφραστικά λάθη. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό λάθος στη μετάφραση που αλλάζει το νόημα εδώ στο κείμενο το δανέζικο. Ε, όσον αφορά το περιεχόμενο της εκθέσεως, νομίζω ότι είναι καλή ιδέα, όπως προανέφερα να προταθεί αυτή η συζήτηση, να διεξαχθεί συζήτηση με το Συμβούλιο, όμως κάποια κομμάτια της διατύπωσης έκθεσης μου δημιουργούν προβλήματα και δεν μπορώ να τα αποδεχτώ. Ίσως να είναι απλώς θέμα ορολογίας, αλλά η διατύπωση στο κείμενο που έχω μπροστά μου μου δημιουργεί δυσκολίες. Στο σημείο 9, Φερρυπίν, λέει ότι εκφράζουμε τη λύπη μας λόγω των δυσκολιών που προέκυψαν με το Συμβούλιο στη διαδικασία της απαλλαγής για τα οικονομικά έτη 2008-2009. Ε, νομίζω ότι είναι ανακριβής διατύπωση. Ε, είναι λόγω δυσ... Δεν είναι λόγω δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε. Πάντα το Συμβούλιο δεν απαντούσε σε ερωτήσεις του Κοινοβουλίου. Ε, είχαν προκύψει κάποια θέματα και το Κοινοβούλιο δεν μπορούσε να αποδεχτεί πλέον την άρνηση να απαντήσει το Συμβούλιο και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα. Μετά στο σημείο 16 λέει ευχαριστεί την Δανική Προεδρία για την υποκοδομητική συμβολή της καθ' τη διάρκεια διαδικασίας απαλλαγής για το 2010. Λυπάται ωστόσο που η Δανική Προεδρία δεν κατόρθωσε να διατηρήσει τα κεκτημένα της Ισπανικής και της Σουηδικής Προεδρίας. Είμαι δανός. Την χάνει να είμαι δανός και δεν έχω αντίρρηση όσον αφορά την έννοια Δανία. Αλλά γιατί να ευχαριστούμε την Δανική Προεδρία. Εντάξει, πράγματι η Δανική Προεδρία ε, ήταν πολύ ευχάριστη απέναντί μας, αλλά πρέπει να πω ότι όσον αφορά την επίτευξη των στόχων, η Δανική Προεδρία ε, απέδωσε, πέτυχε λιγότερους στόχους από τη Ισπανική και από τη Σουηδική Προεδρία και αυτό δεν ήταν λόγο του Συμβουλίου. Η Σουηδική Προεδρία μας έστειλε διάφορες απαντήσεις σε ερωτήσεις μας ατύπως. Η Δανική Προεδρία θα μπορούσε να είχε κάνει το ίδιο. Το Δανικό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους παρότρινε να το κάνουν και δεν το κάνανε τελικά. Οπότε δεν βλέπω γιατί τους ευχαριστούμε. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Δανική Προεδρία ακολούθησε την βασική γραμμή που ακολουθεί πάντα το Συμβούλιο και πέτυχε πολύ λιγότερους στόχους από τη Ισπανική και η Σουηδική. Κρίμα. Και λυπούμε όλος ιδιαίτερος, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Πρέπει να τα διαπιστώνουμε διαφορετικά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δεχόμαστε ένα μοντέλο όπου η Προεδρία μπορεί να είναι απλώς καλή απέναντί μας και να μας χαϊδεύει το κεφαλάκι και εμείς να τους ευχαριστούμε. Ε, μετά, το σημείο 24. Εκεί καλείται η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να προβεί σε διάλογο με το Συμβούλιο. Ε, νομίζω ότι είναι λάθος προσέγγιση. Πάντα θέλουμε διάλογο με το Συμβούλιο. Καλέσαμε το Συμβούλιο σε κάθε συνεδρίασή μας. Το πρόβλημα είναι ότι σε διάφορε περιστάσει και επί ιδανική προεδρία επέλεξε το Συμβούλιο να μην παραστεί. Άρα δεν είναι θέμα του ότι εμεί δεν θέλουμε διάλογο. Πάντα θέλαμε διάλογο και θέλουμε διάλογο. Άρα δεν είναι σωστό ε, να το παρουσιάζουμε έτσι. Να λέμε ότι θα πρέπει να επιδιώκουμε το διάλογο. Το Συμβούλιο θα έπρεπε να δεχτεί ότι επιθυμούμε εμείς το διάλογο, εμφανιζόμενοι όταν προσκαλούνται στην Επιτροπή μας και απαντώντας στις ερωτήσεις που τους βάζουμε. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό να είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι αυτή είναι η διαδικασία. Αλλά αν συμφωνήσουμε να αλλάξουμε αυτά τα σημεία, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση και μπορούμε μετά να συνεχίσουμε τις συζητήσεις με την Κυπριακή Προεδρία επί τη βάση αυτής της, ε, με βάση αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ για αυτές τις παρατηρήσεις και, τις, και τα σχόλιά σας. Ο κύριος Σοντή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, Ινιές που συνεχίζει αυτή τη δύσκολη δουλειά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να έχουμε πλέον το σύνολο των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεσή της και εγώ προσωπικά θέλω να επαναλάβω κάποια ερωτήματα που έχω, κάποια ερωτηματικά μάλλον σε σχέση με τη στάση της Επιτροπής μας που επιμένει να κατακαιρματίζει τις γνωμοδοτήσεις μας επί της απαλλαγής χωρίς να υπάρχει νομική βάση. Δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε αν θα δώσετε το λόγο στο Συμβούλιο. Εγώ θεωρώ ότι η έκθεση αυτή θα έπρεπε να είναι ευκαιρία να εκφραστεί κάθε θεσμικό όργανο, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε πρόκειται για το Συμβούλιο. Γιατί περί αυτού πρόκειται από την αρχή ε, της όλης ιστορίας και μιλάω για πολλά χρόνια πριν, δηλαδή το 2007-2008, Ήδη λοιπόν από τότε είδα τον αγώνα που έδινε η δική μας Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ώστε να επηρεάσει και να πετύχει την απαλλαγή παρατηρώ ότι το νομικό ζήτημα, δηλαδή κατά πόσο ναι ή όχι έχουμε δικαίωμα απαλλαγή, δεν έχει ακόμη ληφθεί μια απόφαση οριστική και αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Νομοθετούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι δίκαιο εφαρμόζεται, τι ισχύει υπάρχει κίνδυνος με, τον κατακαιρματισμό αυτών των χορηγήσεων απαλλαγών. Τι θα πει η Δημοκρατία, θα πει ότι το Κοινοβούλιο ελέγχει, αυτό είναι ο βασικός ρόλος του Κοινοβουλίου, να ελέγχει την εκταλιστική εξουσία. Και στο πλαίσιο του ελέγχου εντάσσεται και η έγκριση ή μη έγκριση των λογαριασμών και της διαχείρισης της εκτελεστικής εξουσίας. Ε, το 2010 είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργήσαμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι δηλαδή η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία, ε, είναι ένα νομικό πρόσωπο, έχει νομική προσωπικότητα πλέον. Έχουμε πλέον μία ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ένα μοναδικό νομικό πρόσωπο. Δεν είναι μια λέσχη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η νομική προσωπικότητα λοιπόν τελικά θα έχει ε, την εξουσία χορήγηση απαλλαγή ή όχι. Σε αυτήν την νομική προσωπικότητα δίνουμε αυτό το δικαίωμα. Και δείχνουμε μέχρι στιγμής να μην έχουμε το πολιτικό σθένος να αρνηθούμε την απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εκπροσωπείται από την εκτελεστική μας εξουσία, που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δει κανεί δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο και την ε, έκθεσή του. Αυτό είναι που μου δημιουργεί όλα αυτά τα ερωτηματικά. Τελευταία φορά ψήφισα την απαλλαγή. Γιατί το ελεγκτικό συνέδριο που είναι αν θέλετε το άλλο χέρι της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού που κρατάει και το πιστόλι που είναι οπλισμένο αν θέλετε ε, εξέφρασε κάποιες απόψεις ε, που δεν ήταν και ιδιαίτερα τιμητικές και για τους υπαλλήλους. Φυσικά και όλοι πάλι πρέπει να είναι στη διάθεση της Επιτροπής μας, ώστε να μπορούμε εμείς ε, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση και του Κοινοβουλίου, γιατί και αυτό ε, σχολιάστηκε στην έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Εγώ προσωπικά εκφράζω πλέον τα ερωτηματικά μου για την προσέγγιση που ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίσως από πολιτικές πλευράς κάποια στιγμή φτάσουμε σε, αυτή την, ε, σε αυτή το διαχωρισμό, ε, τον κατακαιρματισμό των ε, απαλλαγών. Αλλά το Κοινοβούλιο που έχει εξουσία επί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που έχουμε εμείς είναι να έχουμε στο χέρι, αν θέλετε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δώσουμε απαλλαγή ή να μην δώσουμε απλή και να διώξουμε την Επιτροπή με πρόταση μομφή. Αυτή είναι η προβλεπόμενη πολιτική ισορροπία, η προβλεπόμενη από τι συνθήκε. Ε, φυσικά και είναι ατομική βόμβα ε, η πρόταση μομφή, αλλά οι συζητήσει όλε που έχουν γίνει ε, δεν νομίζω ότι έχουν υπόψη τι συνθήκε και το πώ ερμηνεύονται αυτέ. Εκπλήσωμε που σε μια επιστολή λέει η Κομισιόν ότι πρέπει να χωριστεί σε τμήματα η διαδικασία τη απαλλαγή. Μπορεί να του βολεύει αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστή συνθήκη, χωρί να είμαι βέβαιο ότι θα γίνει αυτό. Και επαναλαμβάνω, ζητώ να γίνει μια ανεξάρτητη νομική μελέτη άκρο υψηλού επίπεδου για να δούμε κατά πόσον έχουμε ή όχι δικαίωμα να χορηγούμε απαλλαγή στο Συμβούλιο. Δεν πέρασε η πρόταση αυτή που έκανα, το αίτημά μου και το επαναλαμβάνω. Για να μην υπάρχουν παρανοήσει μεταξύ ημών βουλευτών και των ε, κυβερνήσεων των κρατών που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Οντή. Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει το λόγο. Κύριε Αντρέασεν. Thank you, Chair. I wanted to support... Ευχαριστώ. Υποστηρίζω τον τελευταίο μιλητή. We eh, understand that there is... Πρέπει να καταλάβουμε ότι η απαλλαγή ε, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσωπικότητα δεν είναι νομική όπως είπε ο κ. Σοντή. Είναι νομική προσωπικότητα ε, ε, και έδωσε νομική προσωπικότητα η συνθήκη της Λισαβόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει σε αυτή την οντότητα, στη νέα οντότητα να δώσουμε ε, την απαλλαγή. Υποστηρίζω τα όσα είπε ο συνάδελφός μου, ο κύριος Σταυρακάκης, όπου ζητά διαφάνεια από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Εάν δεν μπορούμε να προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα, τότε δεν παίζουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ειλικρινές και τίμιο και διαφανές. Και όσον αφορά τα όσα είπε ο Δανός συναδέλφος, Συμφωνώ ότι η Δανική Προεδρία δεν έπαιξε ένα πολύ ειλικρινή ρόλο σε αυτό το παιχνίδι. Είμαι στην Επιτροπή Προπολογισμών και νομίζω ότι οι επιδόσεις τους όσον αφορά τον ετήσιο προπολογισμό και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ήταν αρκετά ασαφείς. Όμως επίσης νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πραγματιστές και τώρα εκ νέου αναφερόμαστε στην απαλλαγή για το Συμβούλιο. Όλοι γνωρίζουμε ότι τον Οκτώβριο θα διαπραγματευτούμε τον προϋπολογισμό του επομένου έτους και τον Νοέμβριο θα διαπραγματευόμαστε ή τουλάχιστον θα είμαστε μέσα των διαπραγματεύσεων για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. Έχοντας αυτό υπόψη, ε, νομίζω ότι αυτή η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, αλλά και αυτή η Επιτροπή, έτσι περαιτέρω, ε, έχει υποβαθμιστεί σε κάποιο επίπεδο προσπαθήσαμε να αρνηθούμε ή να αναβάλουμε την αναβολή στο Συμβούλιο και στο τέλος δίνουμε την απαλλαγή διότι έχουμε πρόβλημα με τον προπολογισμό. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια πιο πραγματιστική στάση. Ευχαριστούμε. Είναι κύριος Σκυλακάκης, όχι Σταυρακάκης, όπως είπατε. Ο κύριος Κυλακάκη. Και πραγματικά δεν θέλει μάλλον να τον μπερδεύουν με κάποιον από άλλη ομάδα. Ε, κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει. Θέλει κάποιος να μιλήσει από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο. Ξέρω ότι υπάρχουν εκπρόσωποι του Συμβουλίου, αλλά από ό,τι κατάλαβα σημειώνεται. Θέλει κανείς ε, να πει κάτι. Δίνω το λόγο στην συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου για τα σχόλια. Θα τα λάβω υπόψη. Και βέβαια αν ε, υπάρχουν προτάσεις, ε, ιδέες, ε, είναι ευπρόσδεκτες. Στρέφομαι προς τον κύριο Σκυλακάκη και την ιδέα που εξέφρασε ότι η Κυπριακή Προεδρία Δεν θέλω να αναφέρω προεδρίες ε, που ε, θεωρούμε ότι δεν έχουν ε, πολλές ελπίδες να δώσουν κάποια αποτελέσματα, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν κάποιες προεδρίες για τις οποίες δεν περιμένουμε πολλά, αλλά δίνουν πολλά και άλλες που περιμένουμε πολλά από αυτές δεν, καταφέρουν να ξεπεράσουν κάποιες πιέσεις και δεν αποδίδουν όσο θα έπρεπε. Άρα είμαι ανοιχτή λοιπόν στο να στραφούμε στην Κυπριακή Πρόεδρε για να έχουμε αποτελέσματα έστω και μερικά, και να φτάσουμε στον τελικό, να δώσουμε την τελική μάχη. Φυσικά και μπορούμε να το προσπαθήσουμε. Στον κύριο Σόντεργκατ να πω ότι όπως πάντα εκτιμώ ιδιαίτερα την ανάλυση, επειδή γνωρίζει καλά και το θέμα αυτό. Κατάλαβα τι είπε, ότι δεν πετύχαμε με την Δανική Προεδρία ε, να έχουμε εξέλιξη, παρότι είχε δεσμευτεί ότι θα είναι διαφανής και θα σημειώσει πρόοδο. Αφού λοιπόν δεν το πετύχαμε με τους Δανούς, είναι δύσκολο να το πετύχουμε με τους Κυπρίους, αλλά η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Ποιος ξέρει, εγώ συνεχίζω να ελπίζω όσο ζω. Θα σημείωσε φαντάζομαι και η γραμματεία την ανάγκη να καλέσουμε την Κυπριακή Προεδρία το επαναλαμβάνω και εγώ ότι καλό είναι να καλέσουμε την Κυπριακή Προεδρία όταν θα επανεξετάσουμε αυτό το θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τα τρία συγκεκριμένα σχόλια για κάποια εδάφια της έκθεσης, για το 9, ναι, πράγματι μπορούμε να το βελτιώσουμε. Μπορούμε λοιπόν να διατυπώσουμε από κοινού μια τροπολογία. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημείο 16, έχετε δίκιο κύριε Σόντερκαρτ, αλλά το, το ότι είμαστε ευγενίστε σημαίνει ότι δεν είμαστε και αποφασιστικοί και ντόμπροι στην ε, διατύπωσή μας. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση Άλλο είναι μια Προεδρία που με ελαφρά πηδηματάκια ε, το πέρασε το θέμα έτσι και δεν έκανε τίποτα και άλλο είναι μια άλλη Προεδρία η οποία προσπάθησε να υπερκεράσει τις δυσκολίες. Δεν το πέτυχαν ούτε αυτοί, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το διαχωρισμό. Άλλοι προσπάθησαν, άλλοι δεν προσπάθησαν. Μπορούμε να δούμε ε, το ενδεχόμενο τροποποίησης αυτής της παραγράφου, αλλά εγώ θα ήθελα να φανεί αυτό, ότι δεν το προσπάθησα. Σε ό,τι αφορά τώρα το 24, το σημείο 24, να σας εξηγήσω. Καλεί το Κοινοβούλιο την Επιτροπή Ελέγχου του Υπερπολισμού. Με αυτό τι θέλω. Θέλω να διαφυλάξω το δικαίωμα της Επιτροπής Ελέγχου του Υπερπολισμού να συνεχίσει να εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι διάλογος μεταξύ Συμβουλίου και Κοκομπού είναι, είναι ο διάλογος μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η Κοκομπού ε, μπορεί να επεξεργαστεί το θέμα, το είπε και πρόσφατα του Κοινοβουλίου και είχαμε και ένα σαφές δείγμα χθε. Η Επιτροπή μας τη μία ε, ασκεί ε, μάλλον στη μία φορά τη ασκείται κριτική και την άλλη τη θεωρούν την καλύτερη αν μπορεί η Κοκομπού να έχει κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο πριν μας εξαφανίσουν από το χάρτη, εγώ αυτό λέω. Καλή η Επιτροπή είναι το να συνεχίσει, δηλαδή ουσιαστικά να ασχολείται με αυτό το θέμα. Να διατηρηθεί δηλαδή αυτός ο διάλογο, αυτή η σχέση. Δεν υποχρεώνουμε το Συμβούλιο, δεν το ζητάμε το κάνουμε αυτό αναφορά, αν θέλετε, κάνουμε στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προεπολισμού για να διαφυλάξουμε την δυνατότητα τη Επιτροπή Ελέγχου του Προεπολισμού να εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, για τον κύριο Ντί. Κατανοώ αυτό που είπατε, ότι είναι αόριστη, είναι ασαφή η νομική βάση. Και αυτό δεν γίνεται μόνο αυτή τη φορά, πάντοτε εξαρτάται από την ερμηνεία. Και με πολλέ νομικέ βάσει τη συνθήκη έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Και στην προκειμένη περίπτωση το Συμβούλιο δεν είναι μια δεύτερη βουλή αν θέλετε. Συνομοθετεί, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει από το εθνικό επίπεδο κάποιες φορές. Και είναι πολύ πλοκό όλο αυτό. Να έχουμε μια νομική ε, γνωμοδότηση ψηλοπαίδου, ναι, δεν έχω αντίρρηση, αλλά νομίζω ότι και οι υπηρεσίες οι νομικές εδώ εργάστηκαν με πολύ μεγάλη αφοσίωση, μας έδωσαν ενδιαφέροντα στοιχεία. Η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου βέβαια αντί να εργάζεται υπέρ του Συμβουλίου και των Προεδριών του, νομίζω ότι συχνά δημιουργεί προβλήματα και δεν λύνει ε, αντίθετα τα προβλήματα, αλλά τέλος πάντων. Αυτό το σεμινάριο που θα έχουμε και εκεί θα μπορούμε να συζητήσουμε με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια το ρόλο των θεσμικών οργάνων και να τα συζητήσουμε όλα αυτά πολύ πιο ανοιχτά και αν μπορέσει και το Συμβούλιο να είναι λίγο πιο ρεαλιστικό και να έχει έναν πιο ανοιχτό ειλικρινή διάλογο μαζί μας, ίσως με αυτό το σεμινάριο καταφέρουμε να καταλήξουμε και να δούμε αν χρειάζεται αυτή η νομική ε, γνωμοδότηση ή όχι. Αυτή την ατομική βόμβα ε, που είπατε, ε, δεν είναι η πρώτη φορά που επίσημα αυτή την απειλή. Βέβαια όχι για το Συμβούλιο, για πιο σοβαρά θέματα κατά το παρελθόν. Νομίζω ότι ίσως γιατί είμαι φύση αισιόδοξο ε, άνθρωπος, νομίζω ότι επειδή είναι το μόνο θεσμικό όργανο, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε να ξεπεράσουμε κάποιες επεφυλάξεις ενδιασμού και κάποια έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει. Βλέπω τεράστια δυσπιστία. Υπάρχει μια παράνοια του Συμβουλίου για πολιτική χειραγώγηση λοιπά. Οι διοικητικές θα πάνε στο Συμβουλίο είναι ένα ελάχιστο ποσοστό όπως ξέρετε του προπολογισμού της Ένωσης. Ε, το να καταρρεύσει όλη η απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αυτού μόνο του μικρού ποσοστού δεν νομίζω ότι μας δίνει αξιοπιστία. Πρέπει να προσπαθούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια διέξοδο, μια διμερή λύση με το Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να αναγνωρίσει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, την ασυνανοησία και την ε, έλλειψη εμπιστοσύνης. Και αν αναλύσουμε τον προπολογισμό της Ένωσης, πολύ έτσι θα δούμε ότι το ποσοστό που αντιστοιχεί ε, στο διοικητικό προπολογισμό του ε, Συμβουλίου δεν είναι πια και τόσο σημαντικό το ποσοστό. Άρα δεν νομίζω ότι θα βελτιώνει την κατάσταση. Απέναντι στους πολίτες νομίζω ότι θα χάναμε την αξιοπιστία μας αν ρίχναμε ατομική βόμβα για αυτό το ίσονο σημασίας ζήτημα και δεν τη ρίχνουμε για άλλα πολύ σημαντικότερα ζητήματα. Μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Για το 2010 λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Επαναλαμβάνω στο σεμινάριο μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και φυσικά θα προσπαθήσουμε με την Κυπριακή Προεδρία να έχουμε μια συνεργασία με ανοιχτή σε όλες τις τροπολογίες και σε όλες τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο. Οι τροπολογίες πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Ωραία. Πάμε τώρα στο πρώτο σημείο ε, ζητώ και πάλι ε, συγγνώμη από τον κύριο Κοτούνη, επικεφαλής ε, της ε, γενικής, μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης ε, Γεωργίας. ήμουνα λίγο βιαστικός και σας πιάσα εξαπίνης. σας δίνω τώρα το λόγο για να απαντήσετε σε αυτά που έχει στην ε, γνωμοδότησή της εγγράψει η εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να κάνω μια σύντομη δήλωση για τα σχόλια και τις τροπολογίες της εισηγήτριας. Καταρχάς, να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια για τη συμβολή της σε αυτή τη συζήτηση και για την πρόταση ε, επί των άμεσων πληρωμών που είναι μια από τις προτάσεις μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Να πω εξ αρχής ότι υπάρχει μεγάλη έμφαση στην έκθεση της εισηγήτριας γιατί στην ανάγκη για μεγαλύτερη απλούστευση και για διαφάνεια, όπως επίσης και υπάρχει, δίνεται έμφαση στην ανάγκη μείωσης του διοικητικού φόρτου. Συμμεριζόμαστε πλήρως τις ανησυχίες και αυτούς τους στόχους. Ε, όντως, ε, η προετοιμασία της ΚΑΠ, της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ έγινε με βάση αυτά τα στοιχεία. Όλο λοιπόν το πακέτο συνάδει με αυτούς τους στόχους ε, και η άμεσες πληρωμές του πυλώνα 1 λοιπόν, αλλά και όλα όσα προτείνονται για την ανάπτυξη. Ήταν ε, μια μόνιμη ανησυχία και μέρημνα να διατηρήσουμε με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο και εν ώψη των μελλοντικών προτάσεων. Αυτή η αύξηση της διαφάνειας και της απλούστευσης και η μείωση του διοικητικού φόρτου ε, πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με, τις, με τους στόχους πολιτικής ε, της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Πρέπει να εντάσσεται δηλαδή στο γενικότερο πλαίσιο των γενικών στόχων της ε, Επιτροπής μέσα στα πλαίσια αυτής της μεταρρύθμισης. Επίσης είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν εξετάζουμε την πλευρά της εφαρμογής της μεταρρύθμισης. Είναι κάτι λοιπόν που θα εξετάσουμε κατά την τρέχουσα φάση προετοιμασίας της πρότασης και κατά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αλλά και υπό το φως του τι θα συμβεί ε, κατά τη διάρκεια της φάσης εφαρμογής ε, της μελλοντικής ε, ΚΑΠ. Τούτου λεχθέντος, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν κάποια σημεία που θα ήθελα να σχολιάσω και υπάρχουν και κάποια στοιχεία που εμφανίζονται θετικά στην έκθεση, όπως για παράδειγμα το θέμα των ενεργών γεωργών. Το γεγονός ότι δίνεται έμφαση σε μια πιο στοχευμένη ε, υποστήριξη σε αυτούς τους ε, ε, γεωργούς που έχουν γεωργική δραστηριότητα. Από την άλλη, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη διευκρίνηση για το τι ακριβώς ε, είναι αυτό που θα οδηγήσει σε εξαίρεση των γεωργών από τις άμεσες ε, πληρωμές. Και αυτό είναι κάτι που πάντοτε κοιτούσαμε σε σχέση με αυτούς που έχουν γεωργικές δραστηριότητες. Τώρα για, τα άλλα εργαλεία πολιτικής και εδώ πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης και της επίτευξης των στόχων. Αν δούμε λοιπόν την οικολογική διάσταση, δεν συμμεριζόμαστε την επιλογή ε, της εθελοντικής ε, καταβολής ε, πληρωμών για την οικολογία. Αυτή είναι μια έμεση σύσταση της εισηγήτριας εξετάζοντας το επίπεδο των κυρώσεων που θα περιορίζεται μόνο στις πληρωμές ε, οικολογικής φύσεως εφόσον έχει δοθεί μια εθελούσια ε, διάσταση σε αυτές. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, οι οποίοι πάνε χέρι-χέρι με τις ε, στόχους της γεωργίας. Και πρέπει να γίνει υποχρεωτικό ακριβώς για να διασφαλίσουμε πρώτον ότι το μέγιστο, ο μέγιστος αριθμός γεωργών περιλαμβάνονται σε αυτό το σύστημα και δεύτερον ότι οι τρεις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την οικολογία ε, χρησιμοποιούνται, ισχύουν. Και αν δούμε και άλλα συστήματα υποστήριξης, υπάρχει αυτό το θέμα της μείωσης των ανώτατων ορίων που σχετίζονται με το επίπεδο των πληρωμών ε, που έχουν οι γεωργοί. Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να ε, επιδιώξουμε έτσι ώστε να έχουμε μια πιο στοχευμένη σειρά ε, δικαιούχων. Αν υπάρχει αυτό το, αυτή η μείωση, για άλλη μια φορά θα επικεντρώνουμε τις πληρωμές σε μεγαλύτερες γεωργικές εκτάσεις, οι οποίες ε, από άποψη εισοδήματος χρειάζονται λιγότερο αυτές τις πληρωμές, ενώ θα έπρεπε να γίνεται το αντίθετο. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώς σε αυτούς που χρειάζονται τα χρήματα, γιατί η οικονομία κλίμακος δεν τους επιτρέπει να μπουν στην αγορά τροφίμων. Το ίδιο γίνεται και με τους ε, νεαρούς ε, και μικρούς γεωργούς, Στην περίπτωση των μικρών ε, καλλιεργητών ε, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο σύστημα και αν αυτή είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο έτσι θα μπορούμε να επιτύχουμε μια ισορροπημένη πολιτική, η οποία στοχεύει περισσότερο αυτούς οι οποίοι τι χρειάζονται περισσότερο. Εδώ θα σταματήσω κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Θα απαντήσω με χαρά. μου. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ συγκεκριμένη και ακριβή παρουσίαση. Θέλει κανείς ε, να μιλήσει? Είναι βοηθή της κυρίας Χολμάιερ που έχουν σημειώσει τα σχόλιά σας. 17 Σεπτεμβρίου ε, στις 12 το μεσημέρι είναι η ψηφοφορία. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ε, τελειώνουμε αυτό το σημείο και πάμε στο σημείο 13. Ο κύριος Μούλντερ. Ενδιάμεση έκθεση. Ο κύριος Μούλντερ έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Μπορούμε ε, να μεταφέρουμε αυτό το σημείο στις 17 με 18 Σεπτεμβρίου Δεν έχω κάποιο άλλο σημείο, εκτός αν κάποιος έχει κάτι στα διάφορα. Ωραία. Τότε, το ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη συνεδρία στις 17-18 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος ευχαριστεί τους διερμηνείς. Είναι πάντοτε ωραίο να μπορεί κανείς να τελειώνει νωρίς μια τρίτη πρωί, τόσο κοντά στις διακοπές. Καλές διακοπές